των ερωτήσεων. Η επόμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αύριο 5η 17 Δεκεμβρίου 2009 από τις 9 μέχρι, μέχρι τη 1 και από τις 3 μέχρι τη 5 έχει δημοσιευθεί η μέση διάταξη στο διαδίκτυο τέρμα συνεδρίασης.